και ελπίζω να βάλουμε και την τελευταία ψηφίδα σε αυτό το μοσαϊκό. Ε, ούτως ώστε να έχουμε στεναρούς κανόνες για τη χειραγώγηση της αγοράς και του, τα άτομα που έχουν ε, εμπιστευτικές πληροφορίες. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα ψηφίσουμε ε, γύρω στο μεσημέρι. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η συζήτηση για την έκθεση Δίας μέρα για υπηκόους ε, τρίτων χωρών που πρέπει να κατέχουν θεωρήσεις όταν διέρχονται των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντίας Δεμέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διατρέξαμε μακρά πορεία από τότε που ξεκινήσαμε. Κυρίως θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω <clears throat> για πάρα πολύ ε, φιλόδοξο έργο που υλοποιήθηκε από συναδέλφους ε, και σκιώδες εισηγητές ε, που δείχνει την επαγγελματικότητα και το ιδιαίτερα φιλόδοξο επίπεδο συνεργασίας. Το Συμβούλιο στις διάφορες προεδρίες, την Πολωνική, την Ιδανέζικη, την Κυπριακή, την Λιθουανική, και φυσικά είναι αυτονόητο επίσης να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου και κάνω λόγο φυσικά και για την εξονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Είχαμε πάμπολες ε, συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα, οκτώ τριμερεί ε, διαλόγου, Όλα αυτά αντανακλούν τον περίπλοκο χαρακτήρα αλλά και την ιδιαίτερη σπουδαιότητα αυτή τη έκθεση. Ε, και Ουσιαστικά την 25η Ιουνίου καταφέραμε ευτυχώς να συμφωνήσουμε μεταξύ των ε, ε, ομάδων ΕΛΚΑ, ΑΛΔΕ από κοινού και άλλων ομάδων και της ε, Προεδρίας ε, που στην συνέχεια επικυρώθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο, Συμβούλιο της 28 Ιουνίου. Ευχαριστώ όλους για αυτές τις συμφωνίες και ευχαριστώ και για τις διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις που εμπλουτίζουν, εμπλουτίζουν τη συζήτηση οπωσδήποτε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ευχόμουν να είχαμε υψηλότερα επίπεδα συμπτώσεων απόψεων και συμφωνιών. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την ευαισθησία που καταδείχθηκε στο τέλος και από το Συμβούλιο και από την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου με την τοποθέτηση ότι έχουμε ένα καλό κείμενο. Απόδειξη ήταν η έγκρισή του μεμοφωνία. Η συμφωνία που επετέφθη ενισχύει την πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ένα πλαίσιο δίκαιο και αλληλεγγύης προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών μας. Ο στόχος που έπρεπε να υλοποιηθεί ήταν δύσκολος αλλά καταφέραμε να πετύχουμε να δρομολογηθούν να ε, δράσουμε ε, υπέρ των ευαισθησιών για την ε, διασφάλιση της ισότητας αντιμετώπισης όλων των Ευρωπαίων σε αυτό το πλαίσιο. Όλα αυτά στο δύσκολο πλαίσιο της τήρησης ιδιαίτερα ιδιαίτερων ισορροπιών και ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλήξαμε σε σημαντικούς συμβιβασμούς στα θέματα όπως ε, θεωρήσεις διαβατηρίων ε, όσον αφορά και το χερσαίο πλαίσιο και το ε, πλαίσιο των εναέριων μεταφορών. Καθώς επίσης και για τα πληρώματα πλοίων όσον αφορά επίσης και τις ε, δυνατότητες να, παρέχονται, ε, ή να παρέχεται η προστασία προς τους ετούντες άσυλο και, στη, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των ε, ε, δράσεων ε, βλέπουμε και κάποια σημεία τα οποία είναι παρόλα αυτά πολύ σημαντικά και πρέπει να δίνουν απαντήσεις σε τόσα καθημερινά ζητήματα και προβλήματα που πρέπει να ρυθμίζονται. Καταφέραμε να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας για να εξευρεθεί μια ισορροπή λύση όσον αφορά την αμοιβαιότητα στη δράση μας. Έπρεπε να βρούμε αποτελεσματικά μέσα, αλληλέγγυα μέσα χωρίς να αγνοούμε τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δίνουν αλληλέγγυες λύσεις ε, σε προβλήματα τα οποία αφορούν την ζωή των πολιτών μας. Ε, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ε, κάποιων συναδέλφων για τις επιπτώσεις αυτών των μηχανισμών σε τρίτες χώρες. Όμως πρέπει να προστατέψουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και να αναζητήσουμε προβλήματα, στα προ... λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Άσχετα αν είναι Πολωνοί, Βούλγαροι, Τσέχοι, Κύπροι, Κύπροι αυτή η λύση προβλέπει αυτό το πλαίσιο και αυτές τις δυνατότητες προστατεύοντας τις εξουσίες που δίνει το, η συνθήκη της Λισαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε το οριζόντιο πλαίσιο και τα προβλήματα των κατεντολήν πράξεων και κατεξουσιοδότηση πράξεων. Πρέπει να μελετούμε όμως περίπτωση αναπερίπτωση όλες αυτές ε, τις υποθέσεις. Όλα τα νομικά θέματα μπορεί να τύχουν διαφορετικών ερμηνεών. Όμως ο ένας ή άλλος μηχανισμός εξαρτάται από το νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την απόφαση που θα έχουμε λάβει. Όχι μόνο το κείμενο έχει ε, ομόφωνα γίνει δεκτό από το Συμβούλιο, αλλά έχουμε και την ομόφωνη υποστήριξη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων από το, ε, και τον Ιούλιο από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Βλέποντας αυτό ιστορικά έχουμε το θέμα της ε, συζήτησης που εξελίχθηκε από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου για την αλληλεγγύη, την ισορροπία και τον σεβασμό των εξωτερικών δεσμών και σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας υποβάλλω λοιπόν αυτή τη συμφωνία και ευελπιστώ ότι είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα θα το λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Thank you very much, Mr. Vice President. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία και την ευαισθησία αυτού του φακέλου και των δύο μηχανισμών που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση τροπολογίας. Την αναστολή και την αμοιβαιότητα, που είναι ουσιαστική για να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του κοινού συστήματος θεωρήσεων και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Η Κομισιόν δούλεψε ακούραστα με τι ε, διαδοχικέ προεδρίες και το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό που θα οδηγήσει σε αποτελεσματικό και νομικά ορθό μηχανισμό. Ευχαριστώ ιδίω τον κύριο Ντία Στεμέρα για τι τεράστιε προσπάθειε που έκανε για να φτάσουμε σε συμβιβασμό σε αυτέ τι μακρέ και περίπλοκες διαπραγματεύσει. όπου όμως πριτάνευσε πάντα ε, το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των Προεδριών, το εισηγητή των σχεδόν εισηγητών και τη Κομισιόν. Με μεγάλη χαρά σας λέω ότι ολοκληρώσαμε αυτές τις μακρές διαπραγματεύσεις. Οι δύο μηχανισμοί που είναι τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της τροπολογίας ήταν αναγκαίοι για να έχουμε ένα σύστημα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρηση που να μην είναι πάντα ανοιχτό σε καταχρήσεις και που θα εξασφαλίζει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες την ίση μεταχείριση από τους ε, εταίρους των τρίτων χωρών. Ο μηχανισμός αναστολής ιδίω θα εξασφαλίσει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων με τη γνώση ότι όταν δοθούν ε, καθεστώτα ε, απαλλαγμένα τις θεωρήσεις σε υπηκόους τρίτων χωρών, ε, είναι ένα γενικό μηχανισμό αυτό και δεν θα αφορά τη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Και θα έχουμε και ένα φρένο, ένα μηχανισμό ασφαλείας που μπορεί να ξεκινήσει ούτω ώστε να αποφύγουμε τις παραβιάσεις αυτού του μηχανισμού. Έτσι αυξάνουμε την αξιοπιστία του, του συστήματος θεωρήσεων που έχουμε. Επίσης, η Κομισιόν έχει... δεν είναι σίγουρη για το συμβιβασμό που ε, συζητάμε σήμερα παρά την ικανοποίηση που έχουμε γιατί υπάρχει η, η συμφωνία, είμαστε απογοητευμένοι από τη μορφή που επιλέξαμε για το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το τρέχον κείμενο για αυτού του μηχανισμού, γιατί έχουμε ουσιαστικές αμφιβολίες για την ομιμότητα και αποτελεσματικότητά του. Να σας πω δύο λόγια γιατί. Είναι θέμα αρχής. Οι εκτελεστικές και καταξιοδότηση πράξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να έχουμε και καταξιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις στο ίδιο νομοθετικό κείμενο, αλλά για διαφορετικά είδη μηχανισμών. Εδώ δεν συμβαίνει όμως αυτό. Στο συμβασμό, σε μία περίοδο δύο ετών, οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να λυθεί μέσω εκτελεστικής πράξης. Μετά από δύο χρόνια όμως, η διαδικασία θα περάσει στις κατεξιοδότηση πράξης. Επ' αυτού η Κομισιόν είναι αντίθετη. Επιπλέον, η φύση του μέτρου δεν επιτρέπει τη χρήση των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας αφορά μια συγκεκριμένη χώρα, τον οποίον, της οποίας οι υπήκοοι δεν χρειάζονται θεώρηση για την, ε, να επισκεφτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιβάλλει υποχρεώσει σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέλη της Κομισιόν σημαίνει προσωρινή ε, παράκαμψη του κανονισμού ε, απέναντι σε, αυτή την, σε ό,τι αφορά αυτή την τρίτη χώρα. Πρόκειται μια μεμονωμένη κατάσταση. Μην ξεχνάμε όμως ότι η συνθήκη προβλέπει για τις ε, κατευθυνότητες πράξεις ε, γενική μεταχείριση, γενική εφαρμογή. Επίσης υπάρχει και ένας πολιτικός στόχος, να έχουμε πιο αποτελεσματικό μηχανισμό αμοιβαιότητας και αυτό δεν επιτυγχάνεται. Ο τρέχος συμβιβασμός δεν θα είναι αποτελεσματικός γιατί τα δύο πρώτα χρόνια η Κομισιόν μπορεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις, να άρει το, την υποχρέωση θεωρήσεων για κάποιες κατηγορίες ε, της χώρας, ε, διπλωματικά διαβατήρια ας πούμε και τα λοιπά, μόνο για κάποιους πολίτες της χώρας αυτής. Ε, εν ώψη της δουλειάς που θα γίνει την, την Πέμπτη και την, ε, των περαιτέρω εργασιών του Συμβουλίου θέλω να κάνω την εξής δήλωση ο πλευράς Κομισιόν. Η Κομισιόν καλωσορίζει την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 539 ε, του 2000, της τροποποίησης μάλλον του 539 του 2001 για να αυξηθεί η αξιοπιστία του κοινού συστήματος θεωρήσεων και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Όμως, λυπάται η Κομισιόν που οι αρμοδιότητες που δίδονται στην Κομισιόν για την αναθεώ, τον αθεωρημένο μηχανισμό ε, αμοιβαιότητας είναι κάτι την άποψή τη. όχι συμβατά με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η Κομισιόν επιφυλάσσει το δικαιώματο να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει ε, με βάση τη Συνθήκη, ούτω ώστε να διευκρινιστεί αυτό το σημείο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Τώρα, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, θα δώσω το λόγο στην Βεγονίκ Ματιέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να συγχαρώ θερμά τον κύριο Διασδεμέρα, ο οποίος οδηγεί σε κατάληξη δύο χρόνια διαπραγματεύσεων για την μεταρρύθμιση αυτού του κρίσιμου ζητήματος παρά τις ε, πολλαπλές αλλαγές θέσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Μας επιτρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά την ευρωπαϊκή πολιτική για την θεώρηση των διαβατηρίων. Μέχρι τώρα δεν ήμασταν εξοπλισμένοι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της εξαίρεσης ε, της, από την για τρίτο κράτος. Τώρα μπορούμε συλλογικά να αντιδρούμε σε περίπτωση κράτους ε, τρίτου το οποίο επιβάλλει για ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωση θεώρηση ενώ εμείς το έχουμε απαλλάξει. Άρα μπορούμε να ε, εφαρμόσουμε την αρχή της αμοιβαιότητας που έχει θεμελιώδη σημασία και που σημαίνει μια κοινή ευρωπαϊκή διαχείριση των συνόρων και πίστη στις κοινέ μας δεσμεύσεις. Έχουμε ένα μηχανισμό κατάλληλο που μας επιτρέπει σε περίπτωση ταχείας και ουσιαστικής αύξησης των παράνομων εισόδων από ένα, κράτος μέλος, από ένα τρίτο κράτος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναφέρουμε το σύστημα των θεωρήσεων και επίσης μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα για την προστασία του συστήματος του ασύλου με την αποκατάσταση της υποχρέωσης γιατί η εξαίρεση και ορισμένα δικαιώματα που χορηγούμε είναι βεβαίως. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ λίγο πιο αργά. Σας παρακαλώ λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι δυνατόν να σας παρακολουθήσουμε. Η μεταρρύθμιση λοιπόν μας επιτρέπει μια δίκαιη και ρεαλιστική μεταρρύθμιση του εις των διαβατηρίων για να αποτρέπονται καταχρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Φάιον. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάνουμε λόγο εδώ για ένα, σχέδιο έκθεσης από το οποίο εξαρτάται το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων διαβατηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως απορρίπτουμε αρμοδιότητες που έχουμε ως Ευρωκοινοβούλιο στο θέμα της συναπόφασης. Και είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας, ελεύθερη κίνηση των Ευρωπαίων. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και ένα κενό στο Συμβούλιο και δεν κατανοώ πόσο ο κύριος Διεθεμέρα με τον οποίο συνεργαστήκαμε θετικά λέει όχι τώρα στις κατεξουσιοδότηση ε, πράξη όταν έχουμε αυτές τις οριζόντιες δυνατότητες να περάσουμε ως Ε, υπάρχει ο κίνδυνος που εγκυμονεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός ως πολιτικό μέσο από ευρωπαϊκά κράτη για στόχους ε, πολιτικής εκμετάλλευσης ε, έναντι ατόμων που θα προέρχονται από γειτονικά κράτη σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων όπου η χορήγηση ε, της απαλλαγής θεωρήσεων διαβατηρίων ήταν ένα ορόσημο για αυτά τα κράτη. Τι γίνεται με την πολιτική γειτονία. Ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί σε έκτακτες περιπτώσεις. Τι θα γίνει με τα κράτη της, των Δυτικών Βαλκανίων. Θα είναι πάλι υποχρεωμένα αυτά τα κράτη να ε, υπόκεινται, να υπάγονται σε ένα καθεστώ θεωρήσεων διαβατηρίων. Τι γίνεται με τι δημοκρατικέ αρχέ των δικών μα θεσμικών, θεσμικών οργάνων. Με το ίδιο μα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το ίδιο μπορεί να εφαρμόζεται και με το ε, μέτρο τη αμοιβαιότητα. Όλα αυτά αμφισβητούν τη συμφωνία λοιπόν. Γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τι αρμοδιότητε και δικαιοδοσία μα Και για την εκτέλεση των κατεξουσιοδότηση πράξεων όπω είπε ο επίτροπο, Επιπλέον έχουμε ενώπιόν μα την απειλή μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, δεν διαμορφώνει με απόλυτη σαφήνεια την κατάσταση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το γεγονός. Τι συμβαίνει για παράδειγμα σε σχέση με τις ΗΠΑ ή τον Καναδά με την ε, υποχρέωση εισαγωγής ε, ε, της θέσπισης υποχρέωσης θεωρήσεων διαβατηρίων για έξι κράτη της, για τους <clears throat> πολίτες έξι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει έτσι, δεν νομίζω. Δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει έτσι να διαμορφωθεί το πλαίσιο για το μέλλον παρότι απαιτούνται, επαναλαμβάνω, θεωρήσεις διαβατηρίων για έξι ε, κράτη-μέλη. Είναι ένα μέσο το οποίο ποτέ λοιπόν δεν θα χρησιμοποιηθεί από ό,τι φαίνεται. Συνάδελφοι, απευθύνω έκκληση να καταψηφίσετε αυτή την έκθεση σήμερα και να επιτρέψετε έτσι να περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, σε μια δεύτερη φάση να προστατεύσουμε τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίζονται και κατοχυρώνονται με τη συνθήκη της, Λισαβόνα. Λισαβόνας. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημαντικό θέμα που αφορά άμεσα τους πολίτες μας και την, το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας. Είναι ένα απαραίτητο απαραίτητο στοιχείο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αφορά και πλήττει τους νέους που είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα και που δεν θα έχουν από ό,τι φαίνεται ένα ιδιαίτερα ε, θετικό μέλλον. Είναι αρνητικό αυτό το στοιχείο λοιπόν για τους πολίτες μας, για τη σχέση μας με το Συμβούλιο και για όλη συνολικά της Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ε, γείτονές μας. Έχουμε εξαιρετικές υποχρεώσεις όταν θα έρθει η στιγμή να ψηφίσουμε την Πέμπτη για αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να να λάβουμε μέτρα τα οποία θα είναι μια απειλή. Απειλή για τους πολίτες μας και για την ελευθερία ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Αν υπεψηφίσουμε θα απειληθεί αυτό το δικαίωμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίκστραμ. Ο κ. Σόμπερ για την κυρία Φαγιόν έχει μια ερώτηση. Στα πλαίσια της διαδικασίας της μπλε κάρτας, Κυρία Βίφτσον, περιμένετε λίγο. Δέχεστε, κυρία Φαχών, την ερώτηση. Ναι, αν ναι, ε, κύριο Μπερμάη έρχεται το λόγο. Θα ήθελα να παρακαλώσω την εισηγήτρια να μου απαντήσει δύο ερωτήσεις σχετικές με τα Δυτικά Βαλκάνια. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μιλήσατε για το άνοιγμα των Δυτικών Βαλκανίων, την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων και το καθεξής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχετε υπόψη συγκεκριμένα την κατάσταση στα όμορα κράτη, όπως την πατρίδα μου την Αυστρία, με εκατοντάδες λεωφορεία, τα οποία προερχόμενα από χώρες της, ε, των Δυτικών Βαλκανίων μεταφέρουν ε, υποτιθέμενους τουρίστες στην Αυστρία, αλλά μετά επιστρέφουν άδεια. Και το μεταξύ επιβάτες τους έχουν κάπου εξαφανιστεί. Έχετε υπόψη τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και για τους ε, του πληθυσμούς των περιοχών που πλήττονται. Κυρία Φαγιόν. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Ομπερμαϊ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να δώσω μια εξειδικευμένη απάντηση. Γνωρίζω απόλυτα αυτή την περίπτωση σε σχέση με την τελευταία έκθεση της Frontex για την κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε μεγάλη τύχη που προέρχεστε από την Αυστρία. Μια χώρα που δεν έχει προβλήματα που δεν έχει το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών από τα Δυτικά Βαλκάνια. Εσείς έχετε επαφές με υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Και αληθεύει επιπλέον ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί η ροή των πολιτών που ετούνται άσυλο και μάλιστα ε, χωρίς να έχουν δικαίωμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε εναλλακτικέ δυνατότητες και λύσεις ώστε να επιτρέψουμε οι γείτονέ μας των Δυτικών Βαλκανίων να μπορέσουν να συγκλίνουν προς την πορεία προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ έχει τον λόγο τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι μια σημαντική έκθεση γιατί περιλαμβάνει μια ρήτρα διασφάλισης για την προσωρινή αναστολή α, της εξαίρεσης από την υποχρέωση θεωρήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Θα ήθελα να πω ότι ο βασικός σκοπός είναι ότι παρόλα αυτά ό,τι και να συμβαίνει πρέπει να προχωρήσουμε προς την απελευθεροποίηση του καθεστώτος. Έχουμε το μηχανισμό αμοιβαιότητα, αυξάνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και τα, των χωρών μας και ταυτόχρονα στέλνουμε ένα στεναρό μήνυμα, ηχηρό μήνυμα προς τι τρίτε χώρες ότι θα πρέπει να μεταχειρίζονται όλα τα κρατημέλη τον ίδιο τρόπο σε ό,τι αφορά τι θεωρίε και την απελευθέρωση. Θα θέλαμε να μην χρησιμοποιήσουμε τη συζήτηση για τις κατεξουσιοδότηση πράξης ως πρόσχημα για να απορρίψουμε την συμφωνία και να αποφασίσουμε αυτή τη βδομάδα. Έχουμε κάνει τόση προσπάθεια, τόσες συζητήσεις για να φτάσουμε εδώ. Χρειαζόμαστε αυτή την αυξημένη αλληλεγγύη και πρέπει να την κραδένουμε απέναντι στις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους, η κυρία ο κύριος Τζάντνοκα για τρία λεφτά. Η κυρία Τζάντνοκα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον κύριο Ντίας Τεμέρα, τον εισηγητή μας, για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της ε, μακρόπνοης προσπάθειας που κράτησε δυόμιση χρόνια. Ευχαριστώ τον κύριο Ντίας Τεμέρα για τις ε, προσωπικές προσπάθειες που έκανε για να διατηρήσει τη θέση του Κοινοβουλίου όπως απεικονίστηκε στην ψηφοφορία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων δεν είναι πολύ θετικά για την ομάδα των Πρασίνων. Καταρχάς, υπάρχει ε, μια πρόοδος για την αμοιβαιότητα στις θεωρήσεις. Όλοι θα θυμάστε ότι η αρχική τροπολογία που προτάθηκε από τον κύριο Αλεξάνδρο Άλβαρες, τον καλό μου φίλο αυτόν και υποστηρίχθηκε από τους φιλελεύθερους, από κάποιους κοιόδης και από άλλους συναδελφούς που είναι απόντες από την ομάδα δυστυχώς. Αυτή η τροπολογία λοιπόν ε, σήμαινε σχεδόν αυτόματη επανεισαγωγή ε, θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών όταν βάζουν την υποχρέωση θεώρησης για πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν υποστηρίχθηκε 100%. Τώρα ε, το Συμβούλιο Δήμονα να δεχτεί ένα μηχανισμό σε δύο φάσεις. Και στο τέλος, η Κομισιόν, στο τέλος αυτού του μηχανισμού, η Κομισιόν θα πρέπει να εφαρμόσει την ε, αμοιβαιότητα. Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκειά σας, ε, κύριε Μπαρνιέλα, πρέπει να παραδεχτείτε την πρόοδο. Από την άλλη, είμαστε απογοητευμένοι όμω, με τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την προσωρινή αναστολή της ε, εξαίρεσης της υποχρέωσης θεωρήσεων. Οι πράσινοι δεν θεωρούν ότι η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου μπορεί να είναι κριτήριο για την αναστολή. Οι πήκοοι τρίτων χωρών στο θετικό κατάλογο θα πρέπει να τιμωρηθούν για προσπάθειες υπηκών της ίδιας χώρας να χρησιμοποιήσουν το ατομικό δικαίωμα σε άσυλο παρότι δεν θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και δεν θα πρέπει ε, ο μηχανισμός αναστολής να περάσει μέσα από το, τις εκτελεστικές πράξεις. Αν ε, περνάμε μέσα από τη συναπόφαση, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μπορεί να μπλοκάρει και, ο, και τον προσωρινό όπως και τον μόνιμο μηχανισμό. Και θα πρέπει τα κοινοβουλευτικά δικαιώματα και προνόμια να προστατευτούν. Αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, καταλαβαίνετε ότι η ομάδα μου δεν μπορεί να υποστηρίξει τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Κούε. Ο οποίος Έρνστ. 1,5 λεπτό. Η κυρία Έρνστ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι με αυτόν τον κανονισμό και θα πρέπει να το πούμε ειλικρινά, αλλάζει ο χαρακτήρας ε, των θεωρήσεων διαβατηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι η πολιτική χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων είναι ένα μέσο εκβιασμού, εκβιαστικό μέσο, ιδιαίτερα για τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Αν ενισχύουμε κάτι και θέλουμε να ενισχύσουμε κάτι, είναι το θέμα της αλληλεγγύης σε σχέση με τις, ε, μεταξύ των χωρών μα, Αυστρία, Γερμανία. Ο μηχανισμό αυτό λοιπόν είναι, ας το πούμε αυτό, είναι ένας μηχανισμός και ας το πούμε ειλικρινά που οδηγεί στο τέλος τέλος στα, σύνορα της Σερβίας οι τσιγκάνοι ή όσοι μοιάζουν με τσιγκάνους χωρίς λόγο να τους σταματούν και να τους οδηγούν στην επιστροφή, στο δρόμο της επιστροφής. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Στη Μακεδονία λέει ο ομιλήτρια ότι υπάρχει ένα νομοθέτημα που θέτει η ποινική δίωξη τους ετούντες άσυλο και υπάρχουν και απαγορεύσεις ε, ε ταξιδίων. Αυτή είναι η επίπτωση αυτή τη πολιτική και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Σα ερωτώ, πήγατε σε μια από αυτέ τι χώρε. Εγώ πήγα και είδα στη Σερβία τι γίνεται. Ζούσαν σε μια χωματερή άνθρωποι. Όχι επειδή του αρέσει να ζουν σε χωματερή, οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, αλλά επειδή ε, δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ε, με στοχοθέτηση, με ε, περιορισμό και δίωξη ανθρώπων και δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα τέτοιο κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επομιστεί τα ε, καθήκοντά της και να μην υπεκφεύγει όπως το κάνει σήμερα αυτών των υποχρεώσεων και σε τέτοια θέματα υπάρχουν επεφημίες και λένε ότι χάρη στην πολιτική μας οδηγηθήκαμε σε μια τέτοια καλή κατάσταση. Όμως εμείς πρέπει να απορρίψουμε αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η άλλη εγγεγραμμένη, ο κύριος Κοέλιο, δύο λεφτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε πίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο παρατηρήσεις εδώ. Η πρώτη, για τον μηχανισμό αμοιβαιότητας. Συμφωνώ ότι η απόλυτη αμοιβαιότητα στα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων πρέπει να είναι ο στόχος μας με ένα κράτος μέλος όταν υπάρχει κοινοποίηση σε σχέση με ένα τρίτο κράτος ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανεισδοχής όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν άμεση κοινή απάντηση δίνοντας απάντηση από κοινού σε μια κατάσταση που αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να την χάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικής αντιμετώπισης. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Δεύτερο, το θέμα της επανεισδοχή ή το θέμα της αποκατάστασης ε, ε, των θεωρήσεων διαβατηρίων ή της αναστολής, ε, προσωρινής αναστολής θεωρήσεων διαβατηρίων. Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτός ο μηχανισμός πρέπει να απορρέει σε πολύ συγκεκριμένες έκτακτες περιπτώσεις μόνο όταν υπάρχει σημαντική αύξηση όσον αφορά τον αριθμό των παράνομων μεταναστών που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως θέμα. Ε, συμφωνώ με την προσέγγιση που έγινε σε σχέση με τα ε, εξωτερικά θέματα. Αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να είναι αυτόματος. Συμφωνώ με αυτό. Και συμφωνώ όπως υπογραμμίστηκε πιο πριν ότι η ε, ε, ε, εξαίρεση θεωρήσεων διαβατηρίων είναι μία πτυχή μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Η επανεισαγωγή υποχρεώσεων διαβατηρίων δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό το ευρύτερο συνολικό πλαίσιο και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμερίζομαι αυτό που είπαν οι διάφοροι συνάδελφοι ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερες πληροφορίες και να έχει κάνει περισσότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι όμω ιδιαίτερα ευαίσθητο στα θέματα του συναδέλφου ε, Ντίες Αν δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα ευρύτερο συμβιβασμό, είναι καλύτερο να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα. Είναι σημαντικό να συμμετέχει σε αυτέ τι δυνατότητε πληροφόρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Βέιν Χόλτζερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, μια... ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της συνθήκης της Ξαβώνας ήταν η δημιουργία του χώρου της ελευθερίας, της δικαιοσύνης μαζί με την Οικονομική Νομισματική Ένωση και την Εσωτερική Αγορά. Έτσι λοιπόν, οι βασικές αρχές που προτείνονται ε, από το χώρο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν συζητούμε την τροποποίηση του κανονισμού του 2001. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη θεώρηση του διαβατηρίου αποτελεί ένα ζήτημα που δεν έχει αποκλειστικά εθνικό χαρακτήρα. Ο κοινό χώρος της ελευθερίας δικαιοσύνης και, του, και της ασφάλειας ακολουθεί μια κοινοτική στρατηγική, μια κοινή στρατηγική και γι' αυτό το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον παρακολουθούν από κοινού. Και έτσι και οι, λόγοι, τα μελήματα εσωτερικής πολιτικής έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά βεβαίως, κύριε Βέλτσερ, είδα πολύ προσεκτικά και τα νούμερα. Εγώ νομίζω ότι η ευρωπαϊκή προοπτική ενισχύεται πάνω απ' όλα και ο διάλογος για την Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για μια λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή διάσταση πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ίδιου. Ο εισηγητή, ε, για τον οποίο τρέφω κάθε εκτίμηση για την ε, πολύ ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματο και την επικοδομητική του τοποθέτηση, έχει δυστυχώς ε, προς το τέλος του κειμένου δώσει λιγότερη έμφαση από όσοι θα ήθελα εγώ για την ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό προτείνω ότι θα πρέπει να απορριφθεί η πρότασή του, ώστε να έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση και να ενισχυθεί περισσότερο και η παρουσία και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην συζήτηση αυτή. Ε, Μούλτερ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. όπως και η ομάδα μου, θεωρώ ότι η ελευθερία κυκλοφορίας είναι αγαθό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανοιχτή και προς τα τρίτα κράτη. Βεβαίως, πολλές φορές μπορεί κάτι να πάει στραβά και γι' αυτό πρέπει η νομοθεσία, όπως άλλωστε προτείνεται και τώρα, να έχει και μία ρήτρα αναστολής, η οποία να μας επιτρέπει όταν υπάρχουν προβλήματα να τα αποτρέπουμε, να αποτρέπουμε τις καταχρήσεις. Είναι αυτό σημείο κλειδί για την ομάδα των φιλελευθερών και εμένα προσωπικά. Είναι σημαντικό. Εφόσον μια χώρα παραβιάζει ή αφαιρεί από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάποια δικαιώματα ως προς την δυνατότητα εισόδου στη χώρα αυτή, και εμεί, για λόγου αμοιβαιότητα, να πράττουμε το ίδιο για του δικού τη υπηκόου. Πιστεύουμε ότι οι κατεξουδότητε συμπράξεις θα πρέπει να παραμείνουν ως δυνατότητα, είναι πολύ σημαντικό και ως εκ τούτου μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε την πρόταση του συγητού, τον ευχαριστούμε για τη δουλειά του και ελπίζουμε ότι το κείμενό του θα υιοθετηθεί κατά πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Πίρκερ. Δύο λεφτά. Πρόεδρε. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 είχε υποστηρίξει τότε να υπάρξει η απελευθέρωση από διαβατηρίων για τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τότε το σκέφτηκε πολύ προσεκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάτι πολύ συνετό αποφάσισε. Όταν τώρα διαπιστώνουμε ότι τα αιτήματα ετούντων άσυλο από άτομα από αυτή την περιοχή αυξάνονται και βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ετούντων άσυλο προέρχονται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα η Γερμανία, η Ελβετία, διάφορα κράτη υφίστανται τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί Πρέπει να προσέξουμε όταν έχουμε πληθώρα τέτοιων αιτημάτων που είναι αβάσιμα και ασύστατα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Το πιο σημαντικό μέτρο όπως το βλέπω εγώ και το θεωρώ συνετό και αναγκαίο για την καταπολέμηση της κατάχρησης ε, δικαιώματος αίτησης ασύλου είναι η λήψη απόφασης για μια ρήτρα προστασίας, μια δικλίδα ασφαλείας όταν υπάρχει ξαφνική, απρόβλεπτη αύξηση παρανόμων ή ετούντων άσυλο ασύστατα και ε, χωρίς ε, δικαίωμα ή όταν έχουμε μία ε, μη εφαρμογή ε, συμφωνίας ε, επανεισδοχής. Είναι μία πολύ καλή λοιπόν πρόταση και θα βοηθήσει και δεν θα οδηγήσει σε παράλυση του συστήματος χορήγησης ασύλου αλλά θα επιταχύνει την διαδικασία εξέτασης και χορήγησης ασύλου και αυτό είναι ο στόχος που θέλουμε να επιτελεστεί. Και το χαιρετίζουμε σε δεύτερη αντίδραση το μηχανισμό αμοιβαιότητας που θα εισαχθεί. Αυτό θα οδηγήσει στον να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και μεταξύ των κρατών μελών που θα εκφράζεται έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έντσου, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, καταλαβαίνω τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους συναδέλφους για το θέμα της χρήσης των εκτελεστικών πράξεων ή κατευσιοδότηση πράξεων στους μηχανισμούς αναστολής και αμοιβαιότητα που συμφωνήθηκαν. Σέβομαι, σέβομαι τις ε, απόψεις των συναδέλφων επί των θεμάτων αυτών. Να υπενθυμίσω όμως ότι η συμφωνία που φτάσαμε με το Συμβούλιο έχει το, τη δυνατότητα να θέσει τέρμα σε μια απαράδεκτη κατάσταση α, α, έλλειψης ε, ισότιμης μεταχείρισης που αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες απέναντι στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας θα δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουμε απέναντι στη Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Κύπρο και Κροατία την αλληλεγγύη μας ε, γιατί υφίστανται ε, διακρίσεις απέναντι στην πολιτική ε, θεωρήσεων από Αμερικανούς και Καναδούς. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δεχτούμε εν ονόματι της αρχής της αμοιβαιότητας. Παρακαλώ, δείξτε την αμοιβαιότητά σας και την αλληλεγγύη σας. Ο κύριος Γκάμπριλ για δύο λεπτά. Η κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Αγκουστίν Δίες Δεμέρα, τον συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά του, αλλά και για την ε, στράτευση του σε αυτή διαδικασία από την αρχή της. Έχουμε να κάνουμε με που έχουν ε, κρατήσει αρκετό καιρό. Χάρη στην έκθεση αυτή όμως νομίζω μπορούμε να επικεντρωθούμε στην ουσία των αρχών μας, των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και αυτό λόγο να εκφράσει. Έχουμε έναν ορισμό πλέον ο οποίος μας δίνει και όχι μόνο ε, μια ισχυρή βάση για να προχωρήσουμε και πρέπει να επισημάνουμε ότι πέραν των τεχνικών ε, διατυπώσεων απευθύνουμε και ένα σαφές μήνυμα προς τις τρίτες χώρες και εδώ έχουν θέσει τα ουδέτερα αντικειμενικά κριτήρια και έτσι μπορούν να υλοποιηθούν σωστά. Στο τεχνητικό επίπεδο κάθε ε, θέση σε λειτουργία του μηχανισμού αναστολής θα πρέπει να παρακολουθείτε και βέβαια να γίνεται ανάλυση κατά περίπτωση των συνθεκών γιατί είναι ο μόνος τρόπος αυτός να αντιμετωπίσουμε και την υπέρογγη αύξηση των μεταναστευτικών ροών αλλά και τις αδικίες και ο μηχανισμός αμοιβαιότητας επίσης θα πρέπει να λειτουργήσει ώστε να επιφέρει την επιδιωκόμενη ε, το ειδικόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την αποτελεσματικότητα. Πρέπει και οι ελευθερίες να διαφυλαχθούν αλλά και η ασφάλεια. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική των θεωρήσεων διαβατηρίου με σαφείς όρους και ορισμούς και έτσι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Μόνο έτσι όμως. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή ο οποίος μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε σημαντικά βήματα στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προτασιέβιτς, δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση τελειώνει σε λίγο και δείχνει και έδειξε όμως πόσο δύσκολος είναι ο συμβιβασμός. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το συμβιβασμό. Παρότι ο συνδέσμος αυτός καθεαυτός δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός για όλους. Παρ' όλο αυτό, αξίζει να τον υποστηρίξουμε και να σας πω γιατί. Αμά. Για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, μία από τις μεγαλύτερες, ε, τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών τα ιδανικά του Σέγγεν θα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και να τα προστατεύσουμε και απέναντι στις όποιες καταχρήσεις, βεβαίως. Δεν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να χάσουν την πίστη τους σε αυτά τα ιδανικά. Τώρα, για την είσοδο των, Ευρωπαίων, των, συγγνώμη, των πολιτών υπηκών ε, τρίτων χωρών χωρίς θεώρηση και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα η, συνοδευτικά η αίτηση ασύλου, το βασικό είναι να προστατεύσουμε εδώ τα συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων πολιτών και όχι των γραφειοκρατών. Αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη που βαραίνει τους ώμους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τα βγάλει πέρα, επάξια. Έχει δείξει μέχρι στιγμή ότι είναι ικανή να τα καταφέρει. Τώρα, η εξαίρεση από η προσωρινή εξαίρεση μάλλον α, της απελευθέρωσης του μηχανισμού θεωρήσεων για όσους καταχρώνται αυτό το μηχανισμό είναι πολύ σημαντικό. Οι ανατολικοί εταίροι μας όμως περιμένουν μια κίνηση από πλευράς μας και θα πρέπει να είμαστε πιο γενναιόδοροι. Θα πρέπει να δώσουμε αυτή την εξαίρεση από την υποχρέωση θεωρήσεων σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι μια ανάγκη που έχει καταδειχθεί περίτρανα. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στους ομιλητές που ζήτησαν το λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye. Πίκουλα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα της αμοιβαιότητας για χώρες οι οποίες λαμβάνουν μέτρα περιορισμού στη χορήγηση των θεωρήσεων είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό. Θα πρέπει να δούμε όμως τις πιθανές συνέπειες της εφαρμογής της συγκεκριμένης ρήτρας. η διακοπή της χορήγησης θεωρήσεων μετά, για συγκεκριμένη χώρα μετά από την πολιτική αξιολόγηση της συγκεκριμένης χώρας θα επηρεάσει το πολιτικό και κυρίως το οικονομικό περιβάλλον στη συγκεκριμένη χώρα ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται και για χώρες της λεγόμενης γειτονίας. Ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε λοιπόν την πολιτική την οποία ακολούθησε στη συγκεκριμένη περίπτωση το Βέλγιο, το οποίο αντιμετωπίζει με νέες διαδικασίες αρκετά επιτυχής τους ετούντες άσυλο από οποιαδήποτε χώρα, ιδιαίτερα όμω από τις χώρες οι οποίες είναι δεδηλωμένα υποψήφιες. Είναι καλό να στείλουμε ένα μήνυμα ενθάρρυνσης προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν ότι τα σύνορά μας δεν ανήκουν, δεν είναι αξεπέραστα, αξεπέραστα ούτε είναι σύνορα συμφερόντων. Λούνατσεκ, παρακαλώ. Ähm, Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε και η συνάδελφος ε, ε, Στανόφκα, οι πράσινοι δεν θα υπερψηφίσουν αυτό το πακέτο γιατί δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε πρέπει οπωσδήποτε πλήρως να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, εισηγητής για το κοσφοπέδιο ε, πρέπει να τονίσω ότι οι κάτοικοι του κοσφοπεδίου είναι οι μόνοι που μπορούν να ταξιδέψουν κάτι που είναι μια επιτυχία της ε, διεύρυνσης αλλά κάτι να πω στον συνάδελφο Όστα είπατε ότι εκατοντάδες φορτηγά, ε, συγγνώμη, λεωφορεία έρχονται γεμάτα και επιστρέφουν άδεια. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, αυτό σημαίνει ελευθερία διακίνησης. Μπορούν να έρθουν ε, ε, λεωφορεία ε, και εφόσον έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν μπορούν να ε, επιστρέψουν άδεια. Αυτό σημαίνει ελευθερία μετακίνησης gospodine predsjedniče s obzirom na europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika novih imigracijskih valova u europsko društvo το πρόβλημα οφείλεται στο μικρό επίπεδο, στο χαμηλό επίπεδο ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά μέτρα στα πλαίσια της πολιτικής θεωρήσεων Ένωσης. Αυτό το οποίο έχει σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να διαπιστώσουμε ότι κάθε χώρα έχει το δικό του σύστημα χορήγησης θεωρήσεων γιατί είναι κάτι το οποίο ε, άπτεται φυσικά της προστασίας των πολιτών από τρίτες χώρες όπως επίσης και του επίπεδου ανάπτυξης των διαδικασιών αυτών σε κάθε χώρα. Κάθε χώρα έχει ιστορικές, σαν παράδειγμα, σχέσεις με άλλες χώρες, όπως η Κροατία, η δική μου χώρα, με την Βοσνία Ευζεγοβίνη. Και αυτό επιτρέπει στη χώρα μου να προσυπογράψει μια συμφωνία δίμερη με τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας, έτσι ώστε να εισέρχονται στη χώρα μου χωρίς θεώρηση. Ευχαριστώ. Η ελευθερία διακίνησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγάλη αξία και αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα την απολαμβάνουν όχι μόνο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα αμοιβαιότητα. Γιατί μπορούν μόνο να μπουν ε, μερικοί πολίτες ε, χωρίς θεώρηση αλλά όχι ε, να μπουν οι δικοί μας στη χώρα εκείνη. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, γι' αυτό και θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση με την ανάληψη κάποιων μέτρων. Υπάρχουν ε, και νομικές και πολιτικές δυνατότητες με πιέση στα κράτη-μέλη, ώστε να επαναφέρουν ε, την αμοιβαιότητα στον τομέα αυτό, που είναι ένας πολύ καλός τομέας δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και υπερψηφίζω και υποστηρίζω την έκθεση του κυρίου Μέρα. Ευχαριστώ. Μπεμάια. Κυρία Πρόεδρε, η κυρία Λούνατσεκ ε, δεν θέλει να το καταλάβει, αλλά χιλιάδες ε, κάτοικοι τρίτων χωρών καταχρώνται και το σύστημα θεωρήσεων και το σύστημα ασύλου. Η ρήτρα διαφύλαξης μας επιτρέπει να, να στείλουμε την κατάσταση για να μην γίνει ακόμη χειρότερη και γι' αυτό είναι αναγκαία. Είναι ευθύνη των κρατών μελών. Όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα δεν μπορούμε να περιμένουμε η Κομισιόν να αποφασίσει που χρονοτριβεί τόσο πολύ. Πρέπει να αποφασίσουμε σύντομα, ευέλικτα, να, να προσαρμοστούμε στις ε, ε, νέες συνθήκες μετανάστευσης. Ξέρουμε από το παρελθόν ότι όταν εισέλθουν λαθρομετανάστες στη χώρα είναι πολύ δύσκολο κατόπιν να εκδιωχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λούνατσεκ, υπάρχει μία μπλε κάρτα για σας. Εντάξει, παρακαλώ. Ε, εγώ είμαι η κυρία Λούνατσεκ. Κύριε ε, λέτε ότι χιλιάδες ε, καταχρώνται του δικαιώματος ασύλου. Δεν ισχύει ο αριθμός ε, ε, του μένων άσυλο στην Αυστρία έχει μειωθεί πάρα πολύ και εφόσον θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης τι εννοείται δυστυχώς δεν υπάρχει ένα τέτοιο κοινό σύστημα κάθε χώρα έχει το δικό της δυστυχώς δεν έχουμε κοινή μεταναστευτική πολιτική αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και όχι αυτά τα επιχειρήματα που αναφέρεται πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δυνατότητα ε, μετάβαση από τη μια χώρα στην άλλη. Και όχι αυτά που λέτε εσείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι Όμπερμαϊερ, όχι Λούνατσεκ. Κοιτάξτε, δεν έκανε καμία ερώτηση. Απλώς η συνάδελφος Λούνατσεκ θεωρεί ότι η κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου δεν υπάρχει. Δεν θέλει να το κατανοήσει. Αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Αλλά είναι προφανές και από την έκθεση ότι η κατάχρηση αυτή δημιουργεί πολλές ανησυχίες στους πολίτες. Πρέπει να βρούμε λύση. Το ότι δεν της αρέσει αυτή η λύση το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η θέση της. Εγώ όμως έχω άλλη θέση. Έτσι είναι στη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Μίμητσα. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με τους μηχανισμούς αμοιβαιότητας, εγώ εξήγησα στις ε, προκαταρκτικές μου παρατηρήσεις τις δυσκολίες αυτές. Να σταθώ τώρα στα θετικά αυτής της συμβιβαστικής λύσης και στο ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός διακοπής ο οποίος θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της πολιτικής μας στον τομέα των θεωρήσεων και θα μας δώσει την δυνατότητα καταπολέμησης των καταχρήσεων. Να είστε σίγουροι ότι ο μηχανισμός αυτός θα είναι ο μηχανισμός της τελευταίας στιγμής ή του τελευταίου δυνατού μέτρου που θα ληφθεί και θα εφαρμοστεί εφόσον και μόνο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Το Κοινοβούλιο θα είναι συστηματικά και τακτικά ενημερωμένο για την ε, εφαρμογή των δύο μηχανισμών. Συνειδητοποιώ την σημασία που έχει η διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης στην περιοχή του Σέγγεν και στις γειτονικέ μας χώρες. Το καθεστώς των ελεύθερων θεωρήσεων ήταν μια διαδικασία μακρά και δύσκολη και δεν πρόκειται εμείς να ανατρέψουμε τη διαδικασία αυτή χωρίς να εξετάσουμε προσεπτικά τις συνέπειες. Να αναφερθώ τώρα για την πολιτική μας της θεωρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Καταρχά, ο μηχανισμό διακοπή χορήγηση θεωρήσεων δεν είναι ένα μηχανισμό ο οποίο στοχεύει ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια και στι χώρε του. Είναι μια γενική διαδικασία για όλε οι χώρες για όλε τι χώρε οι οποίε την κάνουν τη ελευθερία στη χορήγηση θεωρήσεων στο σύνολο τη περιοχή Σέγγεν και θα εφαρμοστεί πιθανώς για όλες, ακόμα και για αυτές οι οποίες θα τύχουν του δικαιώματος εξαίρεσης στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια απαιτεί την ειδικότερη μας προσοχή. Αυτό οφείλεται στις επιπτώσεις που έχει η κατάσταση στην περιοχή αυτή, στις διαδικασίες διεύρυνσης και φιλελευθεροποίησης στον τομέα χορήγησης των θεωρήσεων. Αλλά και οφείλεται στο ότι υπάρχει ε, ακόμα ιδιαίτερα υψηλός, αν και μειούμενος προοδευτικά, αριθμός ετούντων άσυλο από πολίτες των χωρών αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμεθα με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και με τα κράτη-μέλη, παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ, προσεκτικά και αναζητούμε λύση. Αυτή στιγμή είναι διαθέσιμος ο μηχανισμός διακοπής, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση ε, μία ή κάποια άλλη χώρα μέλος να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού δεν οδηγεί βέβαια αυτόματα ε, στην, ε, στο να σταματήσει η χορήγηση των ελευθέρων θεωρήσεων. Απαιτούνται περαιτέρω προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ο μηχανισμός και σωστή αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάστασης. Το Κοινοβούλιο θα κρατείται ενήμερο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ευχαριστώ. Διάστε μέρα, ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που εμπλούτησαν με τα σχόλιά τους τη συζήτηση. Και μάλιστα απόδειξη της ε, σημασίας του θέματος είναι ο μεγάλος αριθμός των ομιλητών, 18 που έλαβαν το λόγο για να εκφέρουν με απόλυτα ειλικρινή και δημοκρατικό τρόπο τις απόψεις τους και τους ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή τους και στα θέματα της έκθεσης και όσους υποστήριξαν την έκθεση και όσους διατύπωσαν επιφυλάξεις. Και έχω και μια παρατήρηση και ένα θέμα ουσίας που θα ήθελα να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, κύριε Μίμητσα, ποιος ερμηνεύει την έννοια τη νομιμότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε μία δήλωση. Ε, μάλιστα το γνωρίζαμε και την αναμέναμε. Αλλά δεν συμμεριζόμαστε την ε, νομική σας ε, κρίση και την νομική σας ερμηνεία σε ό,τι αφορά την ε, νομιμότητα ή τη μη νομιμότητα της νομοθετικής πρότασης. Γιατί έχουμε ταυτόχρονα κατεξουδότηση πράξη και εκτελεστικέ πράξει ε, στο ε, περίπλοκο νομικό ζήτημα της αμοιβαιότητα και τη ε, νομιμότητα αυτής. Τώρα, μετά τη δεύτερη σας παρέμβαση, διαπιστώνω ότι έχετε κάποιες επιφυλάξεις. Δεν συμφωνείτε με την έκθεση, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με ένα μόνο. Τι γίνεται με το μηχανισμό της αναστολής. Εσεί αναπτύξατε το μηχανισμό αναστολή με καλύτερο τρόπο και είπατε ότι δεν συμφωνείτε με το μηχανισμό αμοιβαιότητα, ε, τουλάχιστον με τη νομική του διατύπωση. Κύριε Επίτροπε, δεν ακούσαμε τίποτα ελπιδοφόρο από το στόμα σας σε ό,τι αφορά την νομική διασάφηση του ζητήματος. Ε, τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση προς την Επίτροπο που παρακολούθηση με πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και κατάληξη συμφωνία. Αυτό που έκανε ε, ο εισηγητή είναι να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, και κυρίως το διπλωματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όντως, τα Βαλκάνια δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αυτό που έκανε ο εισηγητή, ο υποφαινόμενος, είναι να προτείνει έναν κανονισμό, ένα μηχανισμό αλληλεγγύης ή μια απάντηση στην έλλειψη αλληλεγγύης. Γι' αυτό θα ήθελα να κατακλείδη να αναφέρω έξι ονόματα, πολύ ισχυρά ονόματα. Όταν κατέρτισα την έκθεση αυτό σκεφτόμουν. Τους Κροάτες, τους Κυπρίους, τους Τσέχους, τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και τους Πολωνούς. Αυτούς είχα κατά νου εκπονώντας την έκθεση. Για όλους αυτούς ζητώ αμοιβαιότητα. Για όλους αυτούς ζητώ την αλληλεγγύη. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, θέλετε το λόγο ίσως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, αγαπητέ Σιγητά, να σας πω πολύ ανοιχτά ότι η Επιτροπή είναι ιδιαίτερος υπέρ του μηχανισμού αμοιβαιότητας όπως αναφέρεται στον κανονισμό. Αλλά, αλλά, αυτό με το οποίο δεν συμφωνούμε είναι οι νομικές διαδικασίες για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο μηχανισμός αμοιβαιότητας και ο μηχανισμός αναστολής και γι' αυτόν ισχύει το ίδιο στηρίζεται πλήρως εγκρίνεται πλήρως στα περισσότερα σημεία του στο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο αυτός ο μηχανισμός από μας. Συμφωνώ λοιπόν, κύριε εισηγητά, ότι πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και σας ευχαριστώ και πάλι για τις προσπάθειές σας καθ' όλη τη διάρκεια των μακροχρονίων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη του συμβασμού που επιτύχαμε και ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής και πάλι. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Μίμητσα. Σας ευχαριστώ θερμά για τις διευκρινήσεις σας, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Και σας ευχαριστώ και για την προσπάθεια που καταβάλατε για να συμπαραταχθείτε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είστε σε δύσκολη θέση. Εγώ και οι συνάδελφοι γνωρίζουμε πολύ καλά την έκθεση αυτή. Εσείς κάνατε τεράστια προσπάθεια αντικαθιστώντας την Επιτροπή Μάλστρεμ και εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια αυτή. Αλλά άσχετα με την ανεξαρτησία σας, την δεδομένη ανεξαρτησία του Επιτρόπου, της θέσης του Επιτρόπου, θα έχετε δυσκολίες να εξηγήσετε στη χώρα σας την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχετε πραγματικά σοβαρές πολιτικές δυσκολίες για να υπερασπίσετε αυτή τη θέση. Γι' αυτό και εύχομαι να έχουμε μια σύγκληση των απόψεων, γιατί αυτό που μας χωρίζει είναι η νομική ε, ερμηνεία που υιοθετεί ο εισηγητής για το μηχανισμό αναστολής και το μηχανισμό της αμοιβαιότητας. Μόνο εκεί διαφέρουμε. Commissario vuole mm, intervenire, no? Quindi... Ο Επίτοπος δεν θέλει ξανά το λόγο, συνεπώς η συζήτηση έχει πλέον περατωθεί και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 12.